Γράφειο 2 του ιστορικού κανονισμού υπό την προεδρία του απερχόμενου Προέδρου δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία συζήτηση ε, της οποίας το θέμα δεν σχετίζεται με τον έλεγχο της εντολής ή την ε, εκλογή των Προέδρων. Όλες, ε, όλα τα έγγραφα για την εντολή των βουλευτών ε, θα διαβιβαστούν στην αρμόδια επιτροπή που θα πρέπει να ε, συγκροτηθεί δυνάμει το άρθρο 196 του κανονισμού. Βάσει του άρθρου 3 εδάφιο 2 του ιστορικού κανονισμού όσο δεν έχει γίνει ο έλεγχος της εντολής ή δεν έχει αποφανθεί αρμόδια επιτροπή για αμφισβήτηση ασδήποτη εντολής, ε, ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους οι εκλεγμένοι βουλευτές ε, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει τη δήλωση για το μη ασυμβίβαστο. Σε σχέση με την πράξη τώρα για την εκλογή με άμεση και καθολική ψηφοφορία των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσοι ασκούν καθήκοντα ασυμβίβαστα με την εντολή του βουλευτή δεν μπορούν να εδρεύσουν στο Κοινοβούλιο Όσοι δεν έχουν υπογράψει ακόμη την δήλωση του μία συμβίβαση και ως εκ τούτου δεν έχουν πλήρη δικαιώματα, καλούνται να το πράξουν αμελητή ε, μπροστά στο ημικύκλιο ε, και να υπογράψουν το σχετικό κατάλογο. Ε, εάν δεν τον πράξουν αμέσως δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, προτού προβούμε στην εξέταση του σχεδίου εμερήσιας διάταξης, θα ήθελα να εκφράσω ε, την ευγνωμοσύνη μου και την τιμή ε, που ε, έχω, που μου κάνετε σήμερα ώστε να μπορέσω να προεδρεύσω στην πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκλογή των Προέδρων και Αντιπροέδρων του Σώματος οι ψηφοφόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν την επιθυμία τους για αλλαγή και ελπίζω σε πέντε χρόνια από τώρα να μπορέσουμε να πούμε ότι συμβάλαμε στην οικοδόμηση μιας δικαιότερης Ευρώπης, εγκύτερης στις ανάγκες των πολιτών της. Βάσει του ιστορικού κανονισμού θα προβούμε σήμερα το πρωί στην εκλογή του Πρόεδρου δυνάμει το άρθρο 15 δάφιο 2 του ιστορικού κανονισμού οι υποψηφιότητε για τη θέση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να κατατεθούν με συνενέση των ενδιαφερομένων από μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον από ένα σύνολο 40 βουλευτών. Οι οδηγίε έχουν διανεμηθεί σε όλου του βουλευτέ. Ε, βάσει των κείμενων διατάξεων του κανονισμού έχω λάβει τις εξή υποψηφιότητες για την εκλογή του Προέδρου ο κύριος Καρίμ, η κυρία Λούνατσεκ, ο κύριος Σούλς, ο κύριος Παύλο Ιγκλέσιας ε, οι υποψήφοι μου έχουν κοινοποιήσει ότι αποδέχονται την υποψηφιότητά τους σε βάση το άρθρο 16 εδάφιο 1 του κανονισμού. Σας υπενθυμίζω ότι για την εκλογή στο πρώτο γύρο της ψηφοφορίας ε, θα πρέπει να έχουν την απόλυτη ψηφοφορία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Ε, τα λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη φυσικά κατά την προσμέτρηση των ψήφων πρωτού προβούμε στην εκλογή θα δώσω το λόγο ε, σε όλους τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά για πέντε λεπτά κατά το όριο. Ο κύριος Ιγκλέσιας. Παύλο Ιγκλέσιας. Ευχαριστώ πολύ. Αποτελεί τιμή η ευκαιρία που έχω να σας απευθύνω το λόγο για να σας παρουσιάσω την υποψηφιότητά μου στην Προεδρία του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο αυτό καλείται να εκπροσωπήσει ε, την κυριαρχία της Ευρώπης και κυρίες και κύριοι θα πρέπει να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων που σημαίνει αυτό σήμερα. Το όραμα της Ευρώπης πολλές φορές λύθηκε αλλά ε, κατάφερε κάθε φορά να ξανασυγκωθεί. Περίπου 60 χρόνια η Ευρώπη ε, ξεκίνησε από την αντίσταση των λαών ε, κατά του φασισμού και των στρατοπέδων εξολόθρευσης. Ε, αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν και πολλοί συμπατριώτες μου για τη δημοκρατία στην Ευρώπη και συμμετείχαν σε αυτό τον αγώνα και σε αυτό το όνειρο για δικαιοσύνη. Δεν φαντάζεστε πόσο περήφανος είμαι ως Ισπανός που τα πρώτα άρματα που μπήκαν στο Παρίσι να το απελευθερώσουν ε, είχαν Ισπανούς μαχητές. Σήμερα που η μεσελοδοξία και η ξενοφοβία μας απειλούν θέλω να θυμίσω τη μάχη της Ευρώπης κατά του φασισμού και υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Κυρίες και κύριοι, το καλύτερο που μας ενώνει στην κοινή μας ιστορία mejor de nuestro continente. στην ήπειρό μας λέω ε, σφυριλατήθηκε σε επαναστάσεις που έκαναν το λαό υποκείμενο δικαίου πέρα από ε, μεγαλοκτηματίες, ε, θρησκείες και εξουσίες. Η Ευρώπη ε, θέλει οι πολίτες να είναι ελεύθεροι και όχι δούλοι σε κανέναν. Όχι δούλοι κανενός. Αυτό είναι η δημοκρατία. Γι' αυτό θα πρέπει να σας πω ότι οι λαοί στους οποίους οφείλουμε τις ελευθερίες και τα κοινωνικά δικαιώματα δεν αγωνίστηκαν για μια Ευρώπη όπου ο λαός να ζει με το φόβο της φτώχειας, του αποκλεισμού, της ανεργίας, της απογοήτευσης ανημποριάς απέναντι στην αρρώστια στις ελίτ έχουν ε, υποκληθεί οι κυβερνήσει σε τι ε, χρηματοπιστωτικέ και αυτό είναι απειλή κατά τη ισότητα, τη ελευθερία, της αδελφοσύνη τη κοινή μα ε, ζωή. Η δημιουργία νέων υπερεθνικών οργάνων δεν θα πρέπει να είναι ει βάρο των λαών. Οι πολίτε μα, οι λαοί μα δεν είναι ούτε ανήλικοι ούτε καμία απικία χρέου, κανενό ταμείου. Δεν έχουν αποκτήσει την ελευθερία του για να υποδουλωθούν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτά δεν είναι αφηρημένα, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι σκαθαλώδης η ε, αφέλεια και η ευκολία με την οποία κινούνται εδώ τα λόμπι στην υπηρεσία μεγάλων εταιριών. Ε, οι εκπρόσωποι των πολιτών ε, τελικά γίνονται εκατομμυριούχοι στην υπηρεσία μεγάλων πολυεθνικών. Αυτό είναι κατά της κυριαρχίας των λαών, κατά της δημοκρατίας και καθιστά τους πολιτικούς εκπροσώπους σε κάστα κυρίες και κύριοι, η δημοκρατία στην Ευρώπη έπεσε θύμα εκτροπής αυταρχικής. Στην περιφέρεια της Ευρώπης η κατάσταση είναι τραγική. Οι χώρες μας έχουν γίνει σχεδόν προτεκτοράτα, νέες απικίες, όπου εξουσίες που δυσεξέλεξε εξέλεξε καταστρέφουν τα κοινωνικά δικαιώματα και απειλούν την κοινωνική και πολιτική συνοχή των κοινωνιών μας. Από την Αμερική τη Λατινική Αμερική έχουμε μάθει ότι το εξωτερικό χρέος έχει σχεδιαστεί για να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί και οι χώρες ε, που αναπτύχθηκαν ε, το έπραξαν μετά από σημαντική διαγραφή χρέους, μετά από λογιστικό έλεγχο. Τα ξέρει και η Γερμανία αυτά. Πριν από λίγο καιρό συνέβησαν εκεί, όχι τόσο παλιά. Έχει να κάνει με τη δημοκρατία. Το χρέος σήμερα είναι ένας τρόπος να υποδουλώνουν οι λαοί του Νότου και να λαιλατούνται. Ε, και με ρατσισμό ορισμένοι αποκαλούν αυτές τις χώρες pigs. Αλλά δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν νοείται Ευρώπη χωρίς τους λαούς του Νότου και χωρίς τους λαούς της Ανατολής που επίσης υφίστανται τους σκληρούς κανόνες της Τρόικα που έχει βαλθεί να καταστρέψει την Ευρώπη και να αφήσει ένα ε, πρόσωπο μιζέριας, φτώχειας και βίας. Υπάρχει όμως εναλλακτική λύση στην ε, πολιτική ε, φτωχοποίησης και στη λαιλασία της εξουσίας και της κυριαρχίας. Θα πρέπει να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων και να είμαστε στο επίκεντρο μιας γνήσιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που να σταματήσει την κατηφόρα της αυταρχικότητας της Τρόικας εδώ μας έχουν στείλει οι πολίτες και όχι ε, οι διάφορες συμφωνίες μεταξύ ελίτ. Το κοινοβούλιο δεν είναι ε, χρυσή συνταξιοδότηση ούτε παρηγοριά. Ε, εγώ δεν μιλάω σε ομάδες του Κοινοβουλίου 5-6 ούτε σε κομματικούς μηχανισμούς. Σε πρόσωπο μιλώ, σε βουλευτές, γιατί έχετε ατομική ευθύνη και ένα συμβόλαιο που έχετε υπογράψει με τους λαούς σας. Απευθύνομαι στους δημοκράτες και στις συνειδήσεις σας. Η πρώτη πίστη στην οποία θα πρέπει να υποκληθούμε είναι απέναντι στους πολίτες που μας εξέλεξαν. Αυτοί δεν κυκλοφορούν στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, ούτε στα ξενοδοχεία εδώ γύρω. Αλλά θυμηθείτε, εκείνοι είναι κυρίαρχοι και αργά ή γρήγορα θα σας ζητήσουν το λογαριασμό για το τι κάνατε στο όνομά τους. Και επίσης απευθύνομαι και όλους ιδιαιτέρως στρέφομαι στους ευρωβουλευτές από τις χώρες του Νότου της Ευρώπης. Είδατε τις συνέπειες, τις πραγματικές που έχουν οι πολιτικές που έχει επιβάλει η Τρόικα. Γνωρίζετε ότι οι πολιτικές λιτότητας ναυάγησαν. Οι χώρες μας δεν είναι φτωχές σήμερα είναι πιο φτωχές και με κατεστραμμένες ε, οικονομίες και με πληγωμένες κοινωνίες, με θεσμικά όργανα όπου οργιάζει η έλλειψη αξιοπιστίας και η διαφθορά. Ε, στο χέρι μας είναι να ορθοποδήσουμε και πάλι. Ψηφίστε ως Έλληνες σήμερα, ως Ιρλανδοί, ως Πορτογάλοι, ως Ιταλοί, ως Τσέχοι, ως Πολωνοί, ως Ρουμάνοι, ως Ισπανοί. Τελειώνω αμέσως, Πρόεδρε όχι μόνο για να μπορείτε να δείτε τον κόσμο κατάματα γυρνώντα στη χώρα σας, αλλά γιατί έτσι θα υπερασπιστείτε την Ευρώπη. Ζητώ την ψήφο σας γνωρίζοντας ότι πολλοί δεν συμφωνείτε ε, με αυτή την ομοιρία στην οποία βρίσκεται η δημοκρατία. Ξέρω ότι πολλοί είστε προσιλωμένοι στην ευημερία των λαών σας. Ο πρόεδρος διακόπτη έξω η λιτότητα και ε, η αυταρχικότητα και αυταρχισμός των χρηματοπιστωτικών. Θα σας διακόψω λέει ο πρόεδρος, δεν έχετε πια το λόγο βγήκαν οι λαοί της Ευρώπης, του Νότου της Ευρώπης στον δρόμο για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία. Είπαν φτάνει πια στις πλατείες και θέλω να σας πω ότι είστε η περηφάνεια και η δημοκρατική καρδιά της Ευρώπης. Ο Πρόεδρος διακόπτει. Συγγνώμη, πρέπει να κλείσετε αγαπητέ συνάδελφε. Συνεχίζει ο μιλήτης. Ε, αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι ορθρό, ούτε ε, γίνεται έτσι η διαδικασία. Σας παρακαλώ αγαπητέ συνάδελφε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδελφούς ε, να μην ε, καταχρώνται το χρόνο αγόρευσης. Ε, ούτως ή άλλως τα επόμενα πέντε χρόνια επόμενος πρόεδρος θα σας επαναφέρει στην τάξη. Ο κύριος Καρύμ. Συνάδελφοι, με για να μιλήσω με αίσθηση καθήκοντος. Όπως πολλοί που φτάνετε εδώ για πρώτη φορά, εγώ ήλθα το 2004 με μεγάλη ελπίδα και ε, ενθουσιασμό για την επανένωση της Υπήρου μας μετά από δεκαετίες διχασμού. Σήμερα όμως, συνάδελφοι, αν επιλέξουμε να ακούσουμε, υπάρχει ένα μήνυμα να ακούσουμε. Ένα μήνυμα που απαιτεί από εμάς να αλλάξουμε πορεία. Από ό,τι μου λένε είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα της εκλογής. Έχει ληφθεί συμφωνία ε, ακόμα και πριν ε, πέσει στις κάλπες η πρώτη ψήφος ε, και ότι θα πρέπει όλοι μας να υποκληθούμε στον απόφευκτο Συνάδελφοι, δεν υπάρχει τίποτε πιο ιερό στον κόσμο της δημοκρατικής πολιτικής από το δικαίωμα της ψήφου, το να ε, ρίξουμε την ψήφο μας για αυτά που πιστεύουμε, να εκφράσουμε την επιλογή μας, η οποία θα αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα αυτών που εκλεγήκαμε να υπηρετούμε. Ε, να δώσουμε φωνή ε, σε αγαπημένα ιδεώδη και αρχές. Αυτό όμως μας καλούν ορισμένοι να πράξουμε σήμερα. Τι ε, έχουμε γίνει πλέον εάν ο πρόεδρος του σώματος αυτού ένα αξίωμα που θα πρέπει να ανέρχεται πάνω από οποιαδήποτε ε, κομματικά συμφέροντα και τις πολιτικές φιλοδοξίες περιορίζεται σε ένα αντάλλαγμα, σε ένα πιόνι τελικά, ένα βραβείο, ε, το πλάν D, ε, σε μια πολιτική ζωή όπου το πλάν A, B και C έχει αποτύχει. Μας είπα στις πρόσφατες εκλογές ότι θα είναι διαφορετικά αυτή τη φορά, ότι θα επικρατήσει της μυστικότητας η διαφάνεια, ότι δεν θα είμαστε δεν θα προσπαθήσουμε απλά να διεκπεραιώνουμε κάποια πράγματα. Οι αρχές θα ε, επικρατήσουν. Η ειλικρινής δημοκρατική πολιτική. Δεν θα γίνονται συμφωνίες πίσω από κλειστέ πόρτες, οπισθοδρομικές. Δυστυχώς όμως, ε, ε, λίγες εβδομάδες μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές μας καλούν να δεχθούμε μια πολύ βολική συνένεση, η οποία συμφωνήθηκε πίσω από κλειστέ πόρτε. Πρόκειται για μια ευτελή, φθαρμένη, απονείδηστη εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν δεν είναι αυτό το όραμα με το οποίο θα μπορούσα ποτέ να συμφωνήσω. Είναι μια εντολή να συνεχίσουμε ακριβώς όπως πριν. Να ε, κλείσουμε τα αυτιά μας στα μηνύματα της πλειοψηφίας των ψηφοφόρων, οι οποίοι έμειναν μακριά από την κάλπη. Τα εκατομμύρια επίσης που ένιωσαν ότι πρέπει να διαδηλώσουν, ενώ ο μόνος τρόπος που τους έχει μείνει, ε, στρεφόμενοι στα άκρα όπως είπε ένας πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, δύσκολα μπορεί κανείς να σεβαστεί ένα κοινοβούλιο που δεν σέβεται τον εαυτό του. Εγώ όμως σέβομαι αυτό το κοινοβούλιο, διότι ενσωματώνει πολλές ελπίδες για το μέλλον. Δεν ασχολήθηκα με την πολιτική για να υπερασπιστώ ένα status quo ή για να εξασφαλίσω υψηλά οφήκια για τους λίγους, τις ελίτ. Όχι. Και είμαι και βέβαιος ότι ούτε και εσείς δεν το κάνετε αυτό. Σε όλη μου την πολιτική ζωή έχω ασπαστεί αυτό το όραμα των Ευρωπαίων που συνεργάζονται ε, από κοινού σε ανοιχτού, δημοκρατικού ε, και δίκαιου θεσμού και θεσμικά όργανα και πολλοί από εσά είμαι ότι έχετε το ίδιο όραμα όπου ένα έθνος μόνο δεν διαμορφώνει τα μονοπάτια που θα ακολουθήσουμε, τις προτεραιότητες που θα ακολουθήσουμε, αλλά δίνουμε τις μάχες μας και δεχόμαστε τα αποτελέσματα. Και το είδαμε και μεταξύ των εθνικών ηγετών, που δεν συμφώνησαν όλοι την προηγούμενη εβδομάδα, όμως συνεργάστηκαν και θα συνεργαστούν, όπως πρέπει να κάνουμε και εμείς για να σεβαστούν τις επιθυμίες του εκλογικού σώματος ε, και να ε, φέρουν αυτή την αλλαγή και την ευκαιρία. Βέβαια, έχουμε ελπίδες για το μέλλον, κοινέ μεν, αλλά με διαφορετικές απόψεις πιστεύουμε ότι μπορούν να επιτευχθούν αυτές. Τα θεσμικά μας όργανα όμως δεν θα πρέπει να είναι όμοιρος ή μιας πολιτικής ε, ομάδας ή να είναι ένα αντάλλαγμα ε, για την εξασφάλιση ελέγχου κάπου αλλού. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί το αξιωμά του, το λειτουργήμά του για να εκφράζει προσωπικές απόψεις, να προωθεί τα προσωπικά του συμφέροντα ή να προχωρεί προσωπικά ο ίδιος στα διοδρομία. Το όχι, έχω ένα πιο ευγενές όραμα για το λειτουργήμα του Προέδρου αυτού του σημαντικού θεσμού. Θα πρέπει ο Πρόεδρος να αντικατοπτρίζει την πολυμορφία του σώματος, όπως το Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύει την πολυμορφία των λαών της Ευρώπης. Θα πρέπει να είναι δίκαιο σε όλους, ανοιχτός προς όλους, να δίνει προσοχή σε όλους, να αντιπροσωπεύει το σώμα με αξιοπρέπεια, με τιμή σε όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα τέτοιο πρόεδρο φιλοδοξώ να γίνω. Δεν θέλω να παίξω πολιτικά Θέλω να βελτιώσω τη φήμη, το κύρος ε, του Κοινοβουλίου. Δεν θέλω τα δικά μου συμφέροντα να προωθήσω, θέλω να προωθήσω τα δικά σας συμφέροντα. Δεν θέλω να επανέλθουμε σε πολιτικές και κλεισμένων θυρών και συμφωνιών περασμένων ετών. Θέλω να ε, στραφώ σε όλους τους Ευρωπαίους που προσβλέπουν ε, στο Κοινοβούλιο με ελπίδα για το μέλλον. Αυτό είναι το όνειρο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα όνειρα αυτά όμως θα γίνουν πραγματικότητα μόνο εάν δεν αφήσουμε την αγγελική μας φύση να ιτηθεί από τους πολιτικούς υπολογισμούς τις προσωπικές φιλοδοξίες. Όταν λοιπόν ε, σταθείτε στην κάλπη για να ρίξετε την ψήφο σας σήμερα μόνοι σας απέναντι στα πιστεύω σας και τη συνείδησή σας για τη δημοκρατική σας επιλογή, τι θα επιλέξετε να ψηφίσετε μια συμφωνία και κλεισμένο των θυρών ή μια ανοιχτή διαφανή δημοκρατική Ευρώπη. Ταπεινά ζητώ την υποστήριξή σα για το δικό μου όρομα ενό Προέδρου που θα είναι άξιο αυτού του σώματο και άξιο των λαών τη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω όλους τους νέο εκλεγέντες αλλά και τους επανεκλεγέντες ε, στο σώμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως μας είπε σήμερα το πρωί ένας αυστριακός δημοσιογράφος, ε, που δουλεύει για ένα αυστριακό ραδιόφωνο, ενισχύθηκε το κοινοβούλιο με αυτές τις εκλογές ε, διότι εμείς αναλάβαμε τη διαδικασία για το διορισμό του Πρόεδρου της Επιτροπής και το κοπήραμε από το Συμβούλιο και ως εκ τούτου ενισχύθηκε ο ρόλος μας. Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η νέα δύναμη δεν πρέπει να τεθεί εν κινδύνο ε, λειτουργώντας με λιγότερο δημοκρατικό τρόπο από όσο θα έπρεπε και γι' αυτό το λόγο, συνάδελφοι, εγώ έχω υποβάλει την υποψηφιότητά μου για πρόεδρος. Εγώ στην πολιτική μου ομάδα, όπως και πολλοί άλλοι εδώ, δεν θεωρούμε ότι είναι αποδεκτό να μας πει κάποιο από το Συμβούλιο πριν από 10 ε, ημέρε περίπου, ποιο να ψηφίσουμε για πρόεδρο εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι δική μα επιλογή αυτή. Και η πολιτική μου ομάδα που αρχικά με είχε διορίσει, είχε, είχε υποβάλει την υποψηφιότητά μου για αντιπρόεδρο, ε, ε, μου ζήτησε να καταθέσω την υποψηφιότητά μου για πρόεδρο, ε, διότι περί αυτού πρόκειται. Η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ταυτίζεται με την φωνή των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν είμαστε γραμματέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είμαστε ρετοί εκπρόσωποι του λαού. Ο καθένα από εμά δεν πρέπει να δεχτεί και να επικυρώσει μία συμφωνία που έχουν μαγειρέψει εκ των προτέρων κάποιοι άλλοι. Ο αγώνα για τη δημοκρατία είναι ιδιαίτερα προσφυλέ ζήτημα για μένα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κοινοβούλιο αλλά και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πω τώρα στι τέσσερι γλώσσε που μιλώ ότι η δημοκρατία σημαίνει επιλογή. Δημοκρατία braucht Alternativen. That's why Γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ, αφού σας είπα σε όλες τις γλώσσες που μιλώ ότι πιστεύω και ως Πρόεδρος ε, θα προσπαθήσω να δώσω στους πολίτες ε, μία απάντηση σε σχέση με αυτό που επιθυμούν από τις εκλογές. Θα λήξει η λιτότητα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν μπορεί η γυραιά Ήπειρος να βιώνει ολοένα και εντονότερη φτώχεια, κυρίως στους νέους, ε, όταν οι νέοι δεν θεωρούν ότι είναι πολλά υποσχόμενοι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, την εκλαμβάνουν ως απειλή. Και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να επενδύσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό θα εργαστώ εγώ αν με εκλέξετε. Νέες θέσεις απασχόλησης, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Πέρα από αυτό, χρειαζόμαστε αξιοπιστία εσωτερική. Θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα με τα κτίρια μα, παραδείγματο χάρη, να τα μετατρέψουμε ούτω ώστε να είναι ενεργειακά αποδοτικότερα. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε την διαφάνεια. Έχουμε ένα κώδικα διοντολογίας εδώ στο Κοινοβούλιο που δεν εφαρμόζεται πάντοτε. Θα πρέπει με χάρη στο αποτύπωμα και την ιχνηλασιμότητα να ξέρουμε ποιος επηρεάζει ποιον και να μην επιτρέπουμε σε κανέναν ε, να αγοράζει κάποιο νομοθέτημα ή τουλάχιστον να το προσπαθεί. Για την ενιαία έδρα τώρα, ως βουλευτές θα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς τι χρειαζόμαστε και πού θα εδρεύουμε και όχι το Συμβούλιο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η πλειοψηφία του Συμβουλίου ούτως ή άλλως ε, ψήφισε και αποφάσισε ότι εμείς θα αποφασίσουμε πού θα εδρεύουμε στο μέλλον. Στη συνέχεια θα πρέπει να ε, αντισταθούμε στον λαϊκό ε, στον ε, εθνικισμό και στον εξτρεμισμό. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν υπέρμαχος ανέκαθεν ναι, των ανθρωπίνων βασικών δικαιωμάτων και αυτό θα πρέπει να συνεχίσει. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτήν την τάση ε, της ε, μη ανεκτικότητας ε, και να καταργήσουμε τη διακριτική μεταχείριση ε, για οποιοδήποτε λόγο, λόγω φύλου, λόγω εθνοτικής προέλευσης, και να υπερασπίσουμε τις βασικές αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφασίσουμε για το μέλλον της Ένωσης. Εάν δεν δράσουμε σωστά τώρα, ε, αυτό που θα συμβεί, και θα παραπέμψω τώρα και στο Μουντιάλ, εάν δεν τα καταφέρουμε τώρα, δεν θα έχουμε ούτε... Ούτε παράταση ούτε πέναλτι. Ε, και αυτό είναι το ζήτημα της δημοκρατίας. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ε, κλείσω λέγοντάς σας και θα γυρίσω στα γερμανικά γιατί θα απευθυνθώ στον κύριο Σούλτς. Ο κύριος Σούλτς πριν από λίγο καιρό ήταν στην Αυστριακή Βουλή σε μια συζήτηση παρών για το μέλλον της Ευρώπης. Και ο Μάρτιν Σούλτς εκεί κατήγγειλε ότι πολύ συχνά λέμε ναι μεν αλλά. Δεν μπορούμε να λέμε πάντα καλά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά καλή μεν η δημοκρατία, αλλά καλή η ενοχή, αλλά. Όταν λες αλλά κάθε φορά αρχίζει ο περιορισμός των δικαιωμάτων που είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ πραγματικά το παίρνω σοβαρά, σας πιστεύω, γι' αυτό ε, κατέρχομαι υποψήφια, γιατί η δημοκρατία χρειάζεται και εναλλακτική πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και ελπίζω να με ψηφίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σούλτς. Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είμαστε ένα ιδιαίτερο θεσμικό όργανο 751 βουλευτές σήμερα συνεδριάζουν εδώ και εκπροσωπούν, εμείς εκπροσωπούμε τους λαούς 28 κυρίαρχων κρατών. Είμαστε ένα νομοθετικό σώμα που αποφασίζει νομοθεσία για 507 εκατομμύρια ανθρώπους σε 28 κυρίαρχα κράτη. Αυτό είναι μοναδικό παγκοσμίως. Μόνο το κοινοβούλιο μας είναι πραγματικά μοναδικό και όλος ιδιαίτερο στην ίδια την υπόσταση και τη φύση του, αλλά και ως προς τα καθήκοντά του. Το γεγονός ότι 750 άνδρες και γυναίκες που εκπροσωπούν, αν έχω πληροφορηθεί καλά, περίπου 300 κόμματα και έθνη 28 κυρίαρχων κρατών εδώ στο Κοινοβούλιο. Αυτό το γεγονός και μόνο ότι συνεδριάζουμε από κοινού και συζητούμε και μπορούμε να συζητούμε για το ποιο θα εκλεγεί πρόεδρος του Κοινοβουλίου και μόνο αυτό το γεγονός λέγω κυρίες και κύριοι δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Είναι από τα μεγαλύτερα ιστορικά επιτεύγματα που ε, πέτυχε ουδέποτε ε, αυτή η Ήπειρος και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό και να το θεωρήσουμε βάση για τις εργασίες μας. Όποιος φτάσει στην κορυφή αυτού του θεσμικού οργάνου έχει ένα καθήκον και μία ευθύνη. Ακριβώς ε, από αυτό που σας περιέγραψα μόλις, απορρέει αυτό και θα πρέπει να εργάζεται προς την ευημερία όλων των ανθρώπων και στα 28 κράτη-μέλη. Το πώς θα γίνει αυτό μπορεί να μην μας βρίσκει σύμφωνους και υπάρχουν διάφορα ρεύματα που εκπροσωπούνται εδώ στο Κοινοβούλιο για τον τρόπο δεν συμφωνούμε όλοι. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι εδώ να συνεργαζόμαστε πέρα από σύνορα και πολιτικές ομάδες. Κανείς από μόνος του εδώ ε, δεν έχει την πλειοψηφία. Μπορεί αυτό να μας λυπεί ενδεχομένως, αλλά αυτή είναι η βούληση των ψηφοφόρων, ανδρών και γυναικών. Γι' αυτό η διεθνή συνεργασία που αποτελεί και τη βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, μεταφέρεται εδώ ως συνεργασία πέρα από σύνορα πολιτικών παρατάξεων και κινημάτων. Γι' αυτό η συζήτηση που κάνουμε εδώ είναι πέρα από κόμματα. Στις εκλογές ε, αυτές ε, υπάρχει ελευθερία ψήφου κατά συνείδηση. Δεν υπάρχει καμία κομματική παραταξιακή πειθαρχία. Ο καθένας μπορεί ε, να ψηφίσει όπως θέλει. Το σκοτάδι μέσα στο παραβάν της ε, ψήφου ε, είναι η εγγύηση για την ελευθερία συζήτηση. Τα τελευταία δυόμιση έτη ε, είχα την ευκαιρία να προεδρεύω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ήταν η μεγαλύτερη τιμή σε όλη μου τη ζωή. Θέλω να σας πω ξεκάθαρα τι επιτύχαμε την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο. Ότι δεν υπάρχει πλέον ιεραρχία στα θεσμικά όργανα. Όταν εξελέγην εγώ υπήρχε ακόμα αυτή η ιεραρχία τα μέλη του Συμβουλίου έλεγαν «Ε, καλά το Κοινοβούλιο». Μετά τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλεγε «Ένα είναι το θεσμικό όργανο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου εδώ στο Κοινοβούλιο αυτό το μοναδικό όργανο ουδής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουδής στην ε, ε, Ευρώπη ε, και στα κράτη-μέλη δεν μπορεί να μας παρακάμψει. Είμαστε η πηγή της δημοκρατικής νομιμότητας στην Ευρώπη αυτή η μεγάλη δημοκρατική πρόοδος. ότι η εκτελεστική εξουσία θα πρέπει να απορρέει από τη δημοκρατική κοινοβουλευτική διαδικασία είναι δικό μας επίτευγμα, είναι δικό μας κατόρθωμα και ε, πηγάζει από την ευρωπαϊκή ιστορία και είμαι ιδιαίτερα περήφανης γι' αυτό. Και κατέρχομαι και πάλι υποψήφιος. Και πολλοί συνάδελφοι νεοεκλεγέντες που με βλέπουν εδώ για πρώτη φορά δεν γνωρίζουν τις εμπειρίες που είχαν οι παλαιότεροι συνάδελφοι. Και πολλές καλές και βέβαια οι άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Και είμαι ο τελευταίος που διεκδικώ το αλάθητο. Και εγώ άνθρωπος είμαι με τις ε, αδυναμίες μου και με τα ισχυρά μου. Παρακαλώ να μου κάνετε μια προκαταβολή εμπιστοσύνη τώρα τους νέους και τους παλιούς μια ανανέωση εμπιστοσύνη, για να μπορέσω να προεδρεύσω αξιοπρεπώς με δημοκρατικά ε, ιδανικά ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα προβούμε τώρα στην επιλογή των ψηφολεκτών. Στην κλήρωση των ε, ψηφολεκτών. Δεν υπάρχει συζήτηση για τις ε, δηλώσεις των υποψηφίων. Μπορώ να σας δώσω το λόγο μόνο αν ε, το ζήτημα που θα θίξετε σχετίζεται με την εκλογή του Πρόεδρου. Παρακαλώ. Διαδικαστικό. Ε, για την εναλλακτική για τη Γερμανία, άρθρα 15 και 181 του κανονισμού ζητώ ονομαστική ψηφοφορία. Θα ήθελα να θυμίσω ότι θέλουμε να δείξουμε στους πολίτες ποιος ψηφίζει τον κύριο Σούλτς. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ε, του έχει ε, προσάψει κατάχρηση πόρων, έχει αρνηθεί να δώσει την απαλλαγή ε, πολιτική ομάδα και όχι μία, δύο ή τρεις. Ε, νομίζω παρακαλώ ονομαστική ψηφοφορία για να δουν οι πολίτες Ευρώπης ποιος είναι ο κύριος Σούλτς. Βάση του εσωτερικού κανονισμού είναι μυστική η ψηφοφορία. Όπως έλεγα λοιπόν, θα κληρώσουμε τους 8 ψηφολέκτες. Ονορέβολε Ρέιντα Τζούλια. Ρέιντα Τζούλια. Συμφωνείτε? Κυρία Ρέντα, συμφωνείτε? Συμφωνείτε, πολύ ωραία. Παρακαλείστε να προσέλθετε στο βήμα. Χων Κάρλος Βιτάλ. Είστε παρόν, συμφωνείτε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ελάτε. Ο κύριος Κώστας Χρυσόγωνος, παρακαλώ. Ο κύριος Χρυσόγωνος. No. Yes, I agree. Grazie, venga Παρακαλώ, ελάτε. Onorevole Ferber, Marcus Ferber. Marcus Ferber. Ευχαριστώ. Onorevole Ceballos Bodil. Ceballos Bodil. Prego. Onorevole Petersen Morten Elbeg. Petersen Morten elbeg Bene due. Onorevole Flasikova Benova Monica. Grazie. Della... Onorevole Kirkos Miltiadis. Miltiadis Kirkos. Bene. Ωραία. Θα αρχίσει η ψηφοφορία τώρα. Θα ε, μοιραστούν τα ψηφοδέλτια. Conforme... Και οι φάκελοι. Βάσει των διατάξεων ε, του κανονισμού μας ε, θα προβούμε τώρα στην ψηφοφορία του Προέδρου. Ε, διανέμονται τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι. Θα έπρεπε λοιπόν στη συνέχεια να σημειώσετε να υπογράψετε μάλλον δίπλα στον υποψήφιο της επιλογής σας, να βάλετε ένα σταυρός δίπλα στον υποψήφιο της επιλογής σας μπορείτε να ε, ε, ζητήσετε και νέο ψηφοδέλτιο αν κάνετε λάθος για να μην θεωρηθεί ε, άκυρο. Εάν έχετε βάλει πάνω από ένα σταυρό, θα θεωρηθεί άκυρο το ψηφοδέλτιο. Όσοι θέλουν να μπουν σε καμπίνες υπάρχουν μπροστά στο ημικύκλιο και στη συνέχεια ε, βάσει των αρχικών του ονόματός σας θα ρίξετε το ψηφοδέλτιο στην αντίστοιχη κάλπη. Δεν χρειάζεται ε, να αναφερθώ ονομαστικά στους υποψηφίους. Θα αρχίσει η ψηφοφορία και οι βουλευτές που μετέχουν στην μυστική ψηφοφορία θα ε, καταγραφούν στα πρακτικά και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπογράψετε τον κατάλογο προτού ρίξετε το ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη και ξαναλέω πρέπει να ε, ρίξετε το ψηφοδέλτιο στην ε, κάλπη που αντιστοιχεί στα αρχικά το ονόματό σας. Θα πρέπει να δείξετε και την ταυτότητά σας στους ψηφολέκτες οι οποίοι θα ψηφίσουν στο τέλος, άρχεται η ψηφοφορία.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

Λοιπόν, καλώς. Ε, ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Lo scrutinio è Παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να συγκεντρωθούν στην αίθουσα R1.1 για να προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ψήφων. Διακόπτεται η συνεδρίαση και θα Δείτε πότε θα επαναληφθεί από τις ε, οθόνες, ακούστε και το κουδούνι να χτυπάει. Ευχαριστώ.